Ευχαριστώ συνάδελφοι. Προχωρούμε στις ετολογήσεις ψήφου. Ένα λεπτό στην έκθεση ε, Μαν Μαλίνοφ. Ε, έχουμε τον πρωτομιλητή του κύριο Νέκοφ. Ευχαριστώ. Υποστήριξα την έκθεση για την ε, μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Και αυτό γιατί η έκθεση εστιάζει σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, το Europass το χρησιμοποιούν άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, αλλά όχι άνθρωποι με χαμηλή εξειδικευσή ή ε, λίγες σπουδέ. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο προσβάσιμο αυτό το πλαίσιο. Ανεξαρτήτως οικονομικών, κοινωνικών συνθήκων ο καθένας μας θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στις ε, περιόδους άσκησης της μαθητής Και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Όλοι μας θα πρέπει να ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η απόκτηση εμπειρίας. Αυτό μπορεί να γίνει με τις περιόδους άσκησης και τις μαθητείες που πολλές φορές ε, είναι και ισοδύναμες με μεταπτυχιακό δίπλωμα. Ελπίζω με τις νέες αυτές διατάξεις αυτό να γίνει δυνατόν. Επόμενος, ο κ. Τζαμπάσκι. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγη ησυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ψήφισα υπέρ της πολύ σημαντικής αυτής έκθεσης, διότι χρειάζεται μία επιγραμμική πλατφόρμα για τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες. Με τον εξυγχρονισμό του συστήματος αυτού όλοι οι πολίτες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτή την πύλη, τη διευρυμένη πύλη, αλλά και τους σχετικούς σπόρους. Το νέο εργαλείο απλουστεύεται, βελτιώνει την κινητικότητα στην Ευρώπη. Η προτεραιότητά μας στις διαπραγματεύσεις είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ορατότητα της πλατφόρμας και υψηλά πρότυπα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι σημαντικό για τους συμπολίτε μας να μπορούν να έχουν εύχριστα εργαλεία στη διάθεσή τους ε, για να μπορέσουν να ε, προβάλλουν τις ε, δεξιότητες τους. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ τη έκθεση αυτή. Χαιρετίζω την θεώρηση του πλαισίου Europass για την βελτίωση τη διαφάνεια δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη. Το Europass είναι μια ε, πολύ κορυφαία πρωτοβουλία για τι δεξιότητε επαγγελματικά προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία και η έκθεση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε αυτό το πλαίσιο να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερη κινητικότητα και προ όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η αναθεώρηση του Europass συνοδεύεται από πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα, δηλαδή η συμπερίληψη ε, νέων ε, δεξιοτήτων, όπως ε, ψηφιακών για παράδειγμα, θα μπορούν έτσι οι πολίτες τις υπηρεσίες υπηρεσίες να τις χρησιμοποιούν για να δημιουργούν παραδείγματος χάρη ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια κτλ. Ψήφισα λοιπόν υπέρ αυτή τη έκθεση και ελπίζω να πετύχουμε στους στόχους μας. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Περνάμε στην έκθεση Λα Μασούρο. Ο κύριο Ζάχραντιλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση τη διάβασα και τη βρήκα πολύ αστεία και πολύ ενδιαφέρουσα έγινε λόγος για την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα των Νέων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους νέους μουσικούς, αλλά ακούμε για την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 2014 δεν είχε ε, τα κριτήρια ε, για να χρηματοδοτηθεί. Και ο κύριος Γιούνκερ τώρα το έχει κάνει μεγάλο θέμα και είναι και επιλέξιμη για 600.000 ευρώ το χρόνο. Αστεία πράγματα. Εγώ γελάω. Τι περίεργα προγράμματα καλύπτει αυτός ο τίτλος «Δημιουργική Ευρώπη». Δημιουργικός Juncker είναι, Creative Juncker, όχι Creative Europe. Και αμφιβάλλω πάρα πολύ αν χρειάζεται υποστήριξη αυτό το εγχείρημα και αυτό και το καταψήφισα. Η Πρόεδρος. είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα, Creative Europe, όντως. Ο κύριος Τζαμπάνσκι, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υποστήριξα την έκθεση διότι δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένας ε, φορέας ε, επιλέξουμε σε χρηματοδότηση. Να θυμηθούμε ότι είναι ένας φορέας ο οποίος το 1976 πρώτο δημιουργήθηκε μετά από μια αλλαγή της πολιτικής ε, της ε, Ένωσης για τον ε, πολιτισμό. Θα δημιουργηθεί πλέον μια νέα εποχή για τη δημιουργική Ευρώπη. Αντιμετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες κατά το παρελθόν. Τώρα όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και την ε, πολιτισμική διαφορετικότητα που είναι και χαρακτηριστικό της Ένωσης. Κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την έκθεση αυτή που θέλει να πλουστευθεί το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και για να διαρκέσει στο μέλλον. Η Ορχήστρα των Νέων έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και πρέπει να υπάρξει μια διαφανή ε, υποστήριξη και χρηματοδότηση για να μπορέσει να επιβιώσει η Ορχήστρα των Νέων. Θα πρέπει η νέοι μουσικοί με, σοβαρές, με καλές επιδόσεις να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο. Είναι ε, μια εξαιρετική ευκαιρία για να ε, διδαχθούν οι άνθρωποι την ε, σωστή νοοτροπία του επαγγελματισμού και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Είναι ένα παράδειγμα για ορχήστρες σε όλο τον κόσμο και καμιά ευκαιρία όπως αυτή, καμία ορχήστρα όπως αυτή παγκοσμίως δεν θα δίνει τέτοια ευκαιρία σε νέους Ιρλανδούς μουσικούς με ταλέντο να μπορέσουν να προβληθούν και στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη, πρέπει να το δεχτώ. Ε, και τώρα, έκθεση Λαμασούρ, ο κύριος Ζαχράντιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Τους αποκαλούμενους φορολογικούς παραδείσους. Τι είναι όμως φορολογικός παράδεισος, είναι μια χώρα που βάσει της, ανεξαρτη... της αρχής της, της κυριαρχίας της, της και το κοινοβουλίο της αποφάσισε να έχει φόρο χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι υγιές ο φορολογικός ανταγωνισμός κατά την άποψή μου. Είναι μια κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας και της ανάπτυξης για τα κάτι μελη όλες αυτές οι προσπάθειες να έχουμε κοινέ φορολογικές βάσεις και συντελεστές είναι ε, παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών μελών, στην ε, φορολογική κυριαρχία των κρατών Είναι απλώς η αρχή και από τη φορολογική βάση θα ξεφύγουμε και θα παρέμβουμε απευθείας και σε άλλα πράγματα, ε, Άμεσου φόρου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορώ λοιπόν να το υποστηρίξω. Είναι κάτι που ανοίγει το κόντι τη και είναι επικίνδυνο κατά με. Ευχαριστούμε από την έκθεση, η έκθεση ΤΑΝΚ. Κυρία Άνεμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ε, οικειοποιείται και σφετερίζεται τον εταιρικό φόρο. Ε, στο Βέλγιο εδώ και δεκαετίες έχουμε κίνημα υπέρ της περισσότερης αυτονομίας για τη Φλάνδρα. Ένα φλαμανδικό κίνημα που έχει φτάσει ε, και σε σημείο που η σημερινή κυβέρνηση το έχει πατάξει και το έχει τερματίσει. Και ε, η καρδιά του κινήματος μας ήταν η φορολογική αυτονομία Άρα η Φλάνδρα να μπορεί να έχει καλύτερη οικονομική ανάπτυξη για το φλαμανδικό πληθυσμό. Και εμεί ως φλαμανδικό κίνημα αγωνιζόμαστε να επανακτήσουμε τη φορολογική μας αυτονομία. Και αντί να την πάρουμε από το Βέλγιο, τη δίνουμε στην Ευρώπη. Ενώ 7 εθνικά κοινοβούλια έχουν αντιταχθεί. Είναι σκάνδαλο, δεν είναι καλή λύση. Άλλη λύση θα πρέπει να βρούμε για τα προβλήματά μας. Και ελπίζω πολύ γρήγορα να τερματιστεί αυτή η κατάσταση για την αφόρητη. Ε, έκθεση Βιώτη, ο κύριος Νέκοφ. Πρόεδρε, υποστηρίζω την έκθεση αυτή για τον προπολογισμό του 2019 και τι κατευθυντήριε γραμμέ του, διότι θεωρώ ότι ενώ το Συμβούλιο υποτείνει νέε πολιτικέ προτεραιότητε, οι προτεραιότητε αυτέ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και από νέα κονδύλια. Θα πρέπει να υπάρξουν νέε δεσμεύσει στον προπολογισμό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο δυναμικό των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν εργαζόμαστε σε προγράμματα για τους νέους θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να έχουν επαρκή κονδύλια από τον προπολογισμό της Ένωσης. Αλλά ανταυτού κάθε πρωτοβουλία για τους νέου φαίνεται να χρηματοδοτείται από περικοπές σε άλλα προγράμματα για να μπορέσουμε να βρούμε τα κονδύλια για τους νέους. Προγράμματα μάλιστα που έχουν αποδείξει την αξία τους στον χρόνο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους νέους πολίτες με μια σειρά από νέα προγράμματα, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνεται μόνο μέσω του Erasmus Συν, ούτε αυτό να υποφέρει, που ήταν πολύ επιτυχημένο στα θέματα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ε, περίπτωση της κατάστασης της Συρία, ο Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σύραξη στη Συρία είναι από τις πιο ολέθριες καταστροφές που αντιμετωπίζουμε. Το ψήφισμα αυτό είναι πολύ κρίσιμο, όχι μόνο για τους Σύρους, αλλά για όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη και την ε, ασφάλεια του κόσμου όλου. Όταν αποφασίζουμε ε, στη Συρία και στοχεύουμε στον Άσαντ και το καθεστώς του, ε, φύγουμε μια πολύ εύθραυστη ισορροπία που θα είναι εις βάρος μας. Για το λόγο αυτό καταψήφισα το παρόν ψήφισμα. Με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται, θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλευρά του προβλήματος και όχι στην πλευρά της λύσης. Ας αναρωτηθούμε τι καταφέραμε συγκεκριμένα ε, με τα περιοριστικά μέτρα και τις κυρώσεις απέναντι σε σύρους αξιωματούχους. Πραγματικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στη διπλωματία και πώς μπορούμε να είμαστε ε, πολυμερεί στη διπλωματία μας και χωρίς αποκλεισμού όταν αποκλείουμε Ιράν και Ρωσία. Γι' αυτό καταψήφισα εγώ το παρόν ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ψηφίσαμε για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Οπότε δεν χρειάζεται εδώ επεξήγηση ψήφου. Ολοκληρώνεται η διαδικασία. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καλή σας όρεξη.